συνεδρίες καθώς και τα κείμενα που έχουν εγκριθεί διατίθενται. Έχετε αντιρρήσεις? Όχι. Άρα θεωρούνται εγκεκριμένα τα συνοπτικά πρακτικά. Ο Πρόεδρος έλαβε από το Συμβούλιο